Κυρίε Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση με τη Δημόσια Ακρόαση σε συνεργασία με την Επιτροπή για το Διεθνές Εμπόριο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ έχουν μια μακροχρόνια σχέση που ξεπερνά τον ε, γενικό διεθνή ορισμό για τις εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές, μια εταιρική σχέση για την πρόθεση κοινών αξιών και αρχών, για την παγκόσμια σταθερότητα και για την αμοιβαία μας ε, ευημερία και ε, ασφάλεια. Η σχέση όμως αυτή έχει δοκιμαστεί πρόσφατα λόγω των ε, διαφορετικών απόψεων στην αντιμετώπιση παγκοσμίων θεμάτων και ε, ε, συγκεκριμένων συγκρούσεων όπως τα κλιματικά ή κάποια εμπορικά ζητήματα. Γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει τέσσερις ομιλητές που έχουν διαφορετικές εμπειρίες και ιστορικό καθώς και πείρα που θα συζητήσουν με τα μέλη που βρίσκονται εδώ σήμερα. Η ακρόαση αυτή είναι μια ευκαιρία για να συνεισφέρουμε και ε, ιδέες στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της ΑΦΕΤ για το μέλλον των σχέσεων Ένωσης για προκειμένου να έχουμε την πρώτη ανταλληλή απόψεων αμέσως μετά την ε, ακρόαση την ίδια. Να καλωσορίσω τους προκεκλημένους μας ομιλητές, ε, τον κύριο Γκάρνερ, πρώην ε, Αμερικανό πρέσβη παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τον δόκτορα Κρίστοφ Φον Μάρσαλ, του Ιδρύματος Διτσάιτ και του, του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ της ΗΠΑ, Πολιτείας τον κύριο Τζέρεμι Σαπύρο επίσης, διευθυντή έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Εξωτερικές Σχέσεις και ο, τέσσερι, ο τέταρτος ομιλητής δυστυχώς δεν ήρθε, οπότε έχουμε μόνο τρεις. Θα ξεκινήσει ο κύριος Γκάρντνερ, πρεσβευτά είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν το Νοέμβριο του 2016. Ανυπομονούμε να μας παρουσιάσετε τη δική σας προοπτική και ερμηνεία των ε, σημερινών, της σημερινής κατάστασης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΠΑ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ. Πολλές ώρες έχω περάσει εδώ στην Επιτροπή σας και σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητώντας τη Συμφωνία TTIP και πολλά άλλα θέματα η τριετή μου διπλωματική αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν μόνο δουλειά για μένα, ήταν και μια προσωπική αποστολή, ένα πολύ προσωπικό για μένα θέμα. Και πάντα ένιωθα και συνεχίζω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι φυσικοί εταίροι που θα πρέπει να συνεργαστούν πάνω σε μια σειρά περιφερειακών και παγκοσμίων προκλήσεων. Καμία από αυτέ τι ενώσει ε, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα μόνη τη, χρειαζόμαστε ένα τον άλλον. Μία εβδομάδα πριν ε, ε, τελειώσει η θητεία μου, τον Ιανουάριο του 2017, έδωσα μια συνέντευξη τύπου, στην οποία ήμουν πολύ ειλικρινής και ε, προειδοποίησα σχετικά με τις θέσεις της νέας κυβέρνησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το μετανιώνω αυτό. θεώρησα ότι πολλά διακυβεύονταν για να παραμείνω σιωπηλό και ακόμα το ίδιο πιστεύω. Μερικοί από εσά μπορεί να γνωρίζετε την προσωπική μου ιστορία. Είμαι εγγονός προσφύγων από τον Ιταλικό φασισμό. Ο Μπενίτο Μουσολίνη ήθελε να ξανακάνει σπουδαία την Ιταλία, τελικά όμως κατέστρεψε τη χώρα του και αποφάσισε... Μάλλον ο παππούς μου διαπίστωσε τι γίνεται όταν οι θεσμοί της δημοκρατίας ε, καθώς και τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και ε, το δικαστικό σύστημα υπονομεύονται. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Μαντελέν Όλπραϊτ μας προειδοποίησε όλους ε, ότι θα πρέπει ε, να προσέξουμε τις απειλές προς την δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Και ε, οι σπουδαίοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση των διατλαντικών αξιών μας. Και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα διστάσει να υποστηρίξει τις αξίες αυτές. Ενάμιση χρόνο μετά την ε, έναρξη της ε, κυβερνηση ε, Τραμπ μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ζημιωθεί πολύ σημαντικά και ελπίζουμε προσωρινά. Ο Υπουργό Πομπέο αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πλησιέστερους εταίρους μας στα όσον αφορά τους πιο σημαντικούς μας στόχους στο εξωτερικό. Αυτό το είπε ε, στις 9 Μαΐου με, την, με αφορμή την, ε, την ημέρα της Ευρώπης. Ωραία λόγια αυτά, αλλά ε, αντίκεινται τελείως ε, στις δράσεις της κυβέρνησή του. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απλά όχημα για την ισχύ της Γερμανίας και στόχο έχει μόνο να κερδίσει, να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εμπόριο. Ο Στίβ Μπάνον τώρα έχει αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο. Ο Τζον Μπόλτον όμως, ο νέος σύμβουλος τη Εθνικής Ασφάλειας, είναι ε, πολύ πιθανό να επιβεβαιώσει τις ε, αντιευρωπαϊκές θέσεις ε, του Προέδρου. Και θεωρεί το διεθνές δίκαιο και τους πολυμερείς θεσμούς ε, περιορισμούς στην κυριαρχία της ε, Αμερικής. Ε, δεν, η πολιτική μπορεί να λέει πρώτη η Αμερική, αλλά τα αποτελέσματα είναι μόνη η Αμερική. Η κυβέρνηση αυτή αποκλίνει από μια πολιτική εξικονταετίας και έχω διαπιστώσει τη συνεργασία μας σε εννέα τομείς. Καταρχάς, η φροντίδα του πλανήτη, τα θέματα αλλαγής του κλίματος, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, Καθώ και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση τη διαφθορά σε όλο τον κόσμο. Ε, έχει γίνει σημαντική βλάβη σε όλους αυτούς τους τομείς. Ε, οι προτεραιότητε αυτέ δεν αποτελούν πια προτεραιότητα. Ο δεύτερο τομέα όπου είχαμε τόσο στενή συνεργασία και με τη δική σα Επιτροπή και την Ίντα ήταν οι οικονομικέ μα σχέσει. Ναι, ωραία, δεν τα καταφέραμε με την TTIP. Είχαμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όμω. Ε, είχαμε σημειώσει πρόοδο και σε θέμα προστασία των δεδομένων μετά από 1,5 χρόνο σκληρών διαπραγματεύσεων και επίσης ε, συνεργαστήκαμε πάνω στο ψηφιακό θεματολόγιο. Επίσης, όσον αφορά την ασφάλεια, είχαμε ε, συνεργαστεί στενά σε θέματα ασφάλειας ε, της τη της ενέργειας, πολιτική ασφάλειας, καθώς και συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά μαζί, λοιπόν, και θα πρέπει να προστατεύσουμε του τομεί αυτού στους οποίου είχαμε σημειώσει πρόοδο η απόφαση αποχώρηση από την ε, Πυρηνική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το Ιράν ε, είναι δείγμα της πολλή ζημιά που έχει γίνει. Η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι είναι διμερής η συμφωνία αυτή και μπορεί μονομερός να αποχωρήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείες από αυτήν ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίκιο έχει που επιμένει να διατηρήσει την ε, αμοιβαιότητα των μέτρων. Θα είναι όμως πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, διότι θα είναι δύσκολο να δώσουμε κάποια ωφέλη στο Ιράν τώρα πια. Ε, οι ρήτρες του 1996 απαγορεύουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να συμμορφώνονται με κυρώσεις που σχετίζονται με την Κούβα, το Ιράν και τη Λιβύη. Πρόκειται όμως για ένα ισχυρό και σκληρό νομικό μέσο, διότι οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στις ΗΠΑ. Εγώ είδα από πρώτο χέρι το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει συμπληρωματικά ε, στις δουλειές του ΝΑΤΟ, όχι ανταγωνιστικά. Εγώ συνομίλησα πάρα πολύ με τους στρατηγούς μας που είναι αρμόδιοι για τις ε, αφρικανικές δυνάμεις και διαπίστωσα τι εξαιρετική δουλειά που γίνεται εκεί. Το ΝΑΤΟ εκεί δεν έχει αρμοδιότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να εμπλακούν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν κάνει εξαιρετική δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεχίσει τι επιχειρήσει αυτέ, ε, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι αυτό υπονομεύει το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν συμβαίνει. Παρόλα αυτά τα αρνητικά ε, φαινόμενα, η επιβολή του νόμου παραμένει τομέας όπου μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνεργαστεί με την Europol πολύ αποτελεσματικά σε θέματα όπως είναι το ε, σοβαρό έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, ε, η ε, κακοποίηση παιδιών ε, κλπ. Θέλουμε λοιπόν να μπορούμε να λαμβάνουμε πιο γρήγορα ηλεκτρονικά στοιχεία ένας από τον άλλο από ό,τι στο παρελθόν. Η πράξη cloud επιτρέπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Πολιτειών να υπογράφει συμφωνίες με ξένες κυβερνήσεις για να διευκολυνθεί η αμοιβαία πρόσβαση σε ηλεκτρονικά στοιχεία. Οι κυβερνήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις που σχετίζονται με την δέουσα επιμέλεια, την δέουσα διαδικασία, τον δικαστικό έλεγχο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρώτη τέτοια συμφωνία ε, προβλέπεται ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου και θα ακολουθήσουν και χώρε όπω είναι ο Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ισλανδία και η Ιαπωνία. Εμεί θα θέλαμε να δούμε μια τέτοια συμφωνία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εδώ κάποια πολιτικά προβλήματα, σχεδόν όμω όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, εκφράσει την υποστήριξή του προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στι διαπραγματεύσει στο όνομα των 28, σε λίγο 27 κρατών μελών. Λοιπόν, πολύ σύντομα, οι ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να επιζήσουν μετά από τέσσερα χρόνια κυβέρνησης του Ντόναλτ Τραμπ. Φυσικά και μπορούν. Ε, ο, νομοθετικός διάλογος, ο διατλαντικός νομοθετικός διάλογος ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικός. Θα έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με ομόφρονες συναδέλφους και στα δύο κόμματά μας ε, και ε, επίκεντρο του διαλόγου αυτού είναι η διατήρηση του Privacy Shield, ε, της ε, ασπίδας της ιδιωτικής ζωής και πιθανότατα και διατλαντικού χάρτη για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ε, ε, αμερικανικές επιχειρήσεις, διότι καταλαβαίνουν πόσο ανόητο πράγμα είναι η εμπορική πόλεμη. Είναι ε, πολύ εύκολο να χάσει κανείς σε έναν τέτοιο πόλεμο. Αυτό το καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, θα θέλαμε να δούμε εμβάθυνση των σχέσεων με πολιτείες και πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η αποστολή σας στη Washington κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την εκπαίδευση Αμερικανών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίκιο έχει να πολύ σωστά θα αδράξει την ευκαιρία να υπογράψει νέες διμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες και θα συνεχίσει να στηρίζει τον ΠΟΕ. Πολύ σωστά αρνείστε να διαπραγματευτείτε υπό την ε, απειλή της ε, κάνεις όπλου. Εγώ ε, έχω βρεθεί σε, τέτοιες, σε τέτοια θέση. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνησή μας όπου μπορεί. Κάποια κράτη-μέλη πιστεύουν ότι η ε, κολακία είναι η καλύτερη τακτική, αλλά ε, έχετε σημαντική δύναμη μόχλευσης, ε, μπορείτε να συνεχίσετε να υγείστε με το παράδειγμά σας και το βάρος της ιστορίας βρίσκεται στους ώμους σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάρνερ για τις συμβουλές του. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Κρίστοφον Μάρσαλ, υφηγητής στο γερμανικό Marshall Fund, πολύ γνωστός για τη θέση του ως επικεφαλής διπλωματικός ε, αντιπρόσωπος της Τάγκιος Φίλε και θα μας μιλήσει για τις διαφορετικές επιλογές στη διατλαντική εταιρική σχέση. Πώς θα αποφύγουμε τη συρρήκνωση ποιες είναι οι επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διατλαντική εταιρική σχέση σε ταραχώδεις καιρούς. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Δόκτωρα Φων Μάρσαλ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται. Είμαι η στο Ίδρυμα German Marshall Ζω στην Ουάσιγκτον και ασχολούμαι κυρίως με τα θέματα της Ευρώπης. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη γενικότερα και τι θα έπρεπε να κάνει ειδικότερα η Γερμανία για να διατηρήσει την φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων. Δεν λέω τι θα περίμεναν οι Γερμανοί από τους εταίρους τους και τι δεν θα άρεσε στους Γερμανούς. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αναρωτιέμαι τι περιμένουν οι εταίροι μας από την Γερμανία, τι περιμένουν οι άμεσοι γειτονές μας, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταξιδεύω στη Βρυξέλλες, στη, στη Βαρσοβία, στο Λονδίνο αλλού και μιλάω με όλους τους επικεφαλείς και αρμοδίους. Ζούμε σε καιρούς πολλών κρίσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές αναταραχές που έρχονται από τα εσωτερικά της δύσης. Το Brexit, η εκλογή του πρόεδρου Τραμπ, ε, το ότι λαϊκιστικά κόμματα ανεβαίνουν στην εξουσία συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει μια αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, η Ρωσία γίνεται επιθετική, η Κίνα γίνεται όλο και πιο κυριαρχική, απολυταρχισμός υπάρχει παντού, για παράδειγμα στην Τουρκία. Δεν είναι όμως όλα τα νέα κακά. Από τότε που συνέγραψα την πρότασή μου τον Νοέμβριο του 2016 είχαμε εκλογές στην Αυστρία και στη Γαλλία με θετικές εξελίξεις και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το συγκριτικό πλανέκτημα της δημοκρατίας λειτουργεί, η ικανότητα της αυτοδιόρθωσης. Παρόλο όμως που είχαμε τα αποτελέσματα τα εκλογικά τα θετικά στην Αυστρία και στη Γαλλία, η γενικότερη εικόνα δεν είναι θετική και αντί να περιμένουμε να αυτοδιορθωθεί το δημοκρατικό σύστημα, μήπως θα πρέπει να υιοθετήσουμε πιο ενεργή στάση και να διορθώσουμε μια επικίνδυνη διαδρομή που ακολουθείται τίθεται αυτό το ερώτημα. Τέσσερα είναι οι απαντήσει. Πρώτον, να αναλύσουμε την κατάσταση με ψυχραιμία και όχι με συναισθηματισμό. Να ακούσουμε τους εταίρου, να δούμε τις αδυναμίε, να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε και να αποφύγουμε τις συγκρούσεις που δεν μπορούμε να νικήσουμε σε αυτές. Ήμουν υπέρ της ε, φιλελεύθερης ένομης τάξης πραγμάτων που ε, δημιούργησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν το κλειδί της επιτυχίας για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Η ΗΠΑ μας έδωσαν μια ομπρέλα ασφάλειας για να ανθίσει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και το έπραξαν τότε και έγιναν όλα αυτά και άνθησε και η οικονομία που είναι η βάση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν γίνει ένα πολύ σημαντικό μπλοκ οικονομικής ισχύω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Όμως βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, στην, στη ΣΥΠΑ για την ασφάλειά μας και για να έχουμε εμπορικούς κανόνες σωστούς για να μπορούμε να έχουμε και σωστές εξαγωγές. Όλα αυτά απειλούνται και οι έρχονται από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις και από πολλές εξελίξεις και μία προέλευση ταραχών που δεν περιμέναμε είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος επιβάλλει δασμούς στο αλουμίνιο, στο χάλιβα, με το πρόσχημα ότι είναι απελή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα επιχείρημα που προκαλεί γέλοτα. Απέσυρε τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, από τη Συμφωνία για το Ιράν. Ε, μπλοκάρει τα πράγματα σε επίπεδο ΠΟΕ. Ε, με αυτή την κατάσταση λοιπόν μπορούμε να κάνουμε δύο λάθη. Μπορούμε να υπερεκτιμήσουμε την αναταραχή και μπορούμε και να υποτιμήσουμε την πρόκληση που αυτό σημαίνει για την Ευρώπη. Ο Τραμπ δεν, ε, δεν καταστρέφει τις, ο, τον σύσσωμη τη φιλελευθερία νομή τάξη, αλλά κάποια, κάποια κομμάτια της. Έχουμε κάποια κοινά συμφέροντα, πρέπει να πιέσουμε την Κίνα να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητική ε, διοκτησία το ελεύθερο εμπόριο, να μειώσουμε την ενεργειακή εξάρτηση τη Ευρώπη από τη Ρωσία, να μην διαδώσουμε τα όπλα μαζική καταστροφή να έχουμε σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και στην ε, Αφρική. Αυτά είναι κοινά που έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ. Συμφωνούμε με πάνω σε αυτού του στόχου, από κοινού και δύο μεριέ. έστω και αν διαφωνούμε για τα μέσα επίτευξη αυτών. Κάποιοι ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα φύγει. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τη ΣΥΠΑ. Και τα δύο αυτά επιχειρήματα είναι παραπλανητικά και επικίνδυνα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα φύγει και δεν θα επιτύχει η διαδικασία επιπαραβάση που έχει ξεκινήσει. Μπορεί μάλιστα να επανεκλεγεί το 2020. Δεν θα μετριάσει τι απόψει του και το στυλ τη εκστρατεία του θα το αντιγράψουν και άλλοι πολιτικοί στι ΗΠΑ τη τη του εκστρατεία. Ε, κοιτάζοντας αλλού για παραδείγματα, η Απονία μου τράβηξε την προσοχή. Ο Τραμπ είπε ότι αποσύρεται από την ε, εμπορική συμφωνία με τον Ειρηνικό, με τις χώρες του Ειρηνικού και η Ιαπωνία το δέχθηκε και μέσα σε ένα χρόνο είχε μια συμφωνία με τους 11 άλλους εταίρους της ζώνης του Ειρηνικού ωκεανού, χωρίς τη ΣΥΠΑ. Ε, Νομίζω ότι το δίδαγμα που μπορούμε να αντιλήσουμε είναι ότι δεν είναι καταδικασμένη η φιλελεύθερη ένωμη τάξη πραγμάτων επειδή οι ΙΠΑ σταμάτησαν να τη στηρίζουν. Μπορεί η ένωμη τάξη φιλελεύθερη να υπηζήσει αν μπορέσουν οι υπόλοιποι ηγέτε να την υπερασπιστούν. Τα δύο ερωτήματα που τίθεται είναι τα εξή. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι το αντίστοιχο. Θα συμφωνούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία πάνω στο γεγονό ότι ο Τραμπ δεν είναι αντίπαλο και δεν θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό τη ω εναλλακτική λύση για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ιαπωνία λοιπόν έρχεται και καταλαμβάνει έδαφος εκεί που το αφήνει οι, Ευρωπαϊκή οι το αφήνουν ελεύθερο. Και άρα χειραφετείται στη συμμαχία τη με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν χειραφετείται ενάντια στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε άσκηση πίεσης και μοχλούς πίεσης, εμπορικές συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει αυτού του κανόνε σε μια στιγμή κατά την οποία η ΕΠΑ είναι στο περιθώριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οριστικοποιήσει και ε, συνάψει συμφωνίε με Καναδά, Μεξικό, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, με πολλέ αφρικανικέ χώρε και με τη Μερκοσούρ. Διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση του κανόνε για τον τρόπο χρήση και προστασία δεδομένων, με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αυτά έχουν συνέπεια στη ΣΥΠΑ, έχουν αποτελέσματα. Αμερικανικέ οργανώσει μου ζήτησαν ζήτησαν να λάβουν περισσότερα email βάσει του GDPR, του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμησιακών Καθεστώτων. Ε, Μία πρόκληση που υψώνεται μπροστά μας είναι το εξής, ότι τα κράτη-μέλη δεν συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Όταν στη Βαρσοβία, στο Παρίσι και στο Βερολίνο τους ρωτώ τι πιστεύετε για τον Τραμπ, οι Γερμανοί ε, ε, συχίζονται και θεωρούν ότι τους φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Η Πολωνία λέει δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις, δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα. Η Γαλλία λέει δεν είναι η πρώτη φορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο Αμερικανό πρόεδρο, οπότε δεν έγινε και κάτι. Ε, στο επίκεντρο λοιπόν των διατλαντικών σχέσεων βρίσκεται η ασφάλεια. Ε, ε, για τους Γερμανούς είναι το εμπόριο και οι επενδύσεις. Για τη Γαλλία είναι να παραμείνει η πολυμερής ένωμη τάξη. Δηλαδή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για το ποια είναι τα βασικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εμπειρία να επιτυγχάνει συμφωνίες και ρυθμίσεις και ε, αλλά δεν είναι καλή στο να τα εφαρμόζει μπορεί να καταλήξει συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να θωρακίσει τις επιχειρήσεις από μια εξοεδαφική ε, παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιράν δηλαδή. Για το κράτος δικαίου. Πάρα πολλές χώρες ε, ε, είχαν ερωτηματικά. Σέβεται η Ουγγαρία τις βασικές αρχές, βασικές αρχές και αξίες. Η Γερμανία και η Γαλλία ήταν οι πρώτες που παραβίασαν τους κανόνες για το δημοσιονομικό σύμφωνο και περίμεναν ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες. Και μετά το έκανε η Ελλάδα και η Ιταλία. Ε, τώρα για τη μετανάστευση. Υπάρχουν κανόνες για το πώς θα ε, διαχειριζόμαστε τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Αλλά κάποιοι δεν θέλουν. Το ίδιο στην Ουκρανία. Ε, για πρώτη φορά μέσα σε δεκαετίες οι Ηνωμένε Πολιτείες άφησαν τη διαχείριση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε συμφωνία με τη Ρωσία για την Ουκρανία και δεν μπορεί να την εφαρμόσει. Άρα, πότε επιτέλους θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά τους κανόνες και να μην προβλέπουμε εξαιρέσει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολα τρυπάκια και εύκολες λέξεις, λύσεις και ε, Πολύ συχνά υπάρχει αντίδραση να μην υπάρχουν αρμοδιότητες που να μεταφέρονται στις Βρυξέλλες. Η πρόοδος εξαρτάται από τη βούληση των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύσουν τη διακυβερνητική συνεργασία. Εάν θέλει να μην μειωθεί το κύρος της η Ευρώπη, τότε θα πρέπει να κάνει περισσότερα και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουν προστασία και από τις εγχώριες απειλές και από τις εξωτερικές απειλές και από τις απειλές στην κοινωνικο-οικονομική τους ασφάλεια. Σε μεγάλο βαθμό αυτό συνάδει με τις προσδοκίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια. Άρα λοιπόν ας επικεντρωθούμε στην ασφάλεια έχουμε είναι πολύ μεγάλο ιστορικό πάρα πολλών υποσχέσεων και πάρα πολύ λίγων επιτευγμάτων. Θυμάστε τον πόλεμο στα Βαλκάνια πριν από 20 χρόνια. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει την αιματοχυσία προτού παρέμβουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θυμάστε ότι έχουμε υποσχεθεί να δράσουμε μαζί. Δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι σήμερα. Η χώρα μου, η Γερμανία, βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματο. Υπογράφουμε δεσμεύσει και δεν τι στηρούμε δεν έχουμε το στόχο του 2% του ΝΑΤΟ και η δικαιολογία μας είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε τους Γερμανούς πολίτες που λατρεύουν την ειρήνη να ξοδέψουν περισσότερα πάνω στην άμυνα. Ε, υπογράψαμε την ΠΕΣΚΟ και λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τους Γερμανούς που αγαπούν την Ευρώπη να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα. Ε, επομένως, θέλουμε να τους ευχαριστούμε όλους με, στα, με τα ωραία λόγια. Και μετά τις συνομιλίες στο Παρίσι και στη Βαρσοβία, είδα ότι πια δεν γινόμαστε πιστικοί. Ε, το Παρίσι έχει την αίσθηση του επίγοντος. Το Βερολίνο όχι. Το Βερολίνο λέει ότι όλα καλά πάνε. Οι αναταραχές κάπου αλλού συμβαίνουν γιατί να αλλάξουμε εμείς εδώ στη Γερμανία. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι πολιτικοί στη Γερμανία και οι τεχνοκράτες αναγνωρίζουν ότι πράγματι οι Γερμανοί πρέπει να κάνουν παραπάνω. Αλλά ποιο θα το πει αυτό στους ψηφοφόρους οι εταίροι δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν γερμανικές δικαιολογίες και έχουν δίκιο. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να πιστεί το γερμανικό κοινό. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις σε όλη τη Γερμανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ο κόσμος είναι έτοιμος να ακούσει. Το πρόβλημα είναι με την ηγεσία με τους ηγέτες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να μην είστε υπερβολικά ευγενικοί με τους ομολόγους σας στη Γερμανία. Προκαλέστε τους. Η Γερμανία πρέπει να αλλάξει γιατί ο πλούτος και η επιρροή συνοδεύονται πάντοτε από την ευθύνη και πρέπει κανείς να την αναλαμβάνει αυτή, να μην παίρνει μόνο το πρώτο κομμάτι. Ιδαλλιώς η σημασία μας ως χώρας αλλά και ως Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βαίνει συρρυκνούμενη σε βάθος χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φον Μάρσαλ. Και τώρα τρίτος ομιλητής, ο κύριος Σαπυρό, Διευθυντής Μελετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα μας μιλήσετε για τις σχέσεις ιπα Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Έχετε το λόγο κύριε Σαπυρό. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας και στο ακροατήριο αυτό. Εάν προσπαθείτε να κατανοήσετε την, την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι προηγουμένως πρέπει να κάνουμε κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις για την την κυβέρνηση. Για να κάνουμε τη σωστή ερμηνεία. Πρώτον, η κυβέρνηση Τραμπ συνολικά δεν έχει καμία στην πραγματικότητα προσέγγιση συγκεκριμένα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη. Ε, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που την αποσχολούν ε, περιστρέφονται όλα γύρω από το εμπόριο και τη μετανάστευση. Δεν εννοώ με αυτό ότι η κυβέρνηση είναι διχασμένη. Ε, είναι ή ότι είναι αυτή η κανονική κατάσταση της Αμερικανικής κυβέρνησης στην πραγματικότητα. Δεν μπορούν να σχηματίσουν μια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής για τα θέματα αυτά. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ο ίδιος ο πρόεδρος, η προσωπικότητά του, η ε, ιδιοσυγκρασία του και η κριτική του ικανότητα δεν δίνει καμία αξία ε, και δεν έχει καμία συνέπεια, αγνοεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και παρεμβαίνει τελείως ε, ξαφνικά και βία χωρίς να έχει προετοιμάσει καθόλου το έδαφος. Αυτό για τους πιο ε, συνετούς και προσεκτικούς συμβούλους του κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που ο καθένα θα επέκρινε κοιτάζοντα την εξωτερική του πολιτική. Κανεί δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τι θα κάνει η κυβέρνηση του Τραμπ για την εξωτερική πολιτική. Ακόμη και αν αυτό το πρόσωπο που προσπαθούσε να μαντέψει ήταν ο ίδιο ο Τραμπ. Ο βασικό τομέα όπου υπάρχει κάποια σχετική συνέπεια και συνοχή στην κυβέρνηση Τραμπ, εξαιρέσει υπάρχουν και εδώ, ήταν το θέμα του διεθνού εμπορίου. Αυτό είναι το ζήτημα που τον έφερε στην πολιτική στη δεκαετία του 80. Ε, Πιστεύει εδώ και 30 χρόνια ότι οι, Ευρωπα... ότι οι έχουν πληγεί από το σύστημα διεθνούς εμπορίου και ότι είναι κακή συμφωνία ε, αυτή που έχουν πετύχει οι Ηνωμένε Πολιτείε χάνοντας χρήματα. Και αυτό επειδή πήραν μέρο στι πολυμερεί εμπορικέ διαπραγματεύσει. Ότι αυτό εμπόδισε τη είπα, να βαρύνουν ε, με την τεράστια οικονομία του όσο έπρεπε στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπε και ο κ. Γκάρντνερ, είναι μια πολυμερή συνωμοσία για να πάρει από τα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών ε, επιτυχεί εμπορικέ συμφωνίε. Και πιστεύει ο κύριο Τραμπ ότι αυτό πετυχαίνει. Επίση, τρίτον, είναι ότι ο κύριο Τραμπ γνωρίζει πολύ λίγα και ε, ε, ενδιαφέρεται πολύ λίγο για την Ευρω... Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη περισσότερο. Δεν τον απασχολεί η άποψη του κατεστημένου ότι όπω πίστευαν οι Αμερικανοί, οι πρόεδροι από τη δεκαετία του 40, η Αμερική θα ωφεληθεί, οι ΕΕ θα ωφεληθούν από τη σταθερότητα και την οικονομική ευημερία των ε, ευρωπαϊκών κρατών. Ο Τραμπ έχει δώσει βάρο στι σχέσεις με την Κίνα και ως προς την Ιαπωνία ε, γεωπολιτικά τον έχουν απασχολήσει πάλι εμπορικέ σχέσει και έχει κοιτάξει μόνο το Μεσανατολή, το Ιράκ και τη Συρία. Ε, ασχολείται με τα μαθήματα ε, εδώ τον ενδιαφέρει να ξεκινήσει κύκλο μαθημάτων γκολφ στην Ιρλανδία. Τόσα ξέρει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήξερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ε, αρμοδιότητα εκ μέρου των κατομελών τη να διπλωματεύεται εμπορικέ συμφωνίε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Και στι τρει πρώτε συναντήσει με εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Τραμπ προσπαθούσε να ε, ε, το καταλάβει, γιατί το εξηγούσε υπεύθυνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολύ ανθεκτικό στην μάθηση ο κύριο Τραμπ. Ε, τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τις σχέσεις ΕΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επί τη κυβέρνηση Τραμπ. Εδώ το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι ξεχάσετε τη στρατηγική Τραμπ για τα θέματα αυτά. Ε, αντισταθείτε στον πειρασμό να δημιουργήσετε μια τεράστια, ένα τεράστιο αφήγημα για την φοβερή αυτή προσέγγιση που θα έχει ο Τραμπ ε, στι σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι ε, διαβεβαιώσει και να σα προσφέρουν οι χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι, δεν θα υπάρχει καμία βεβαιότητα για τη στρατηγική προσέγγιση στον ΗΠΑ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πάντοτε παραλυκόμενο άλλων ε, θεμάτων, όπω εμπορικέ σχέσει με την Κίνα ή ακόμα χειρότερα η διάθεση του Πρόεδρου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η ιδέα που έχει κυκλοφορήσει πολύ και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη και ισχύει ότι οι ενήλικοι ε, που βρίσκονται στην ίδια με τον Τραμπ, ε, η Συμβουλή του, το Κογκρέσο, τα δικαστήρια μπορούν να δημιουργήσουν μια συνεκτική εξωτερική πολιτική προς, τις, ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε άλλο. Αλλά αυτό δεν επιβίωσε στους 15 πρώτους μήνες κυβέρνησης Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε αντίθεση με άλλους Αμερικανούς προέδρους ε, στο Περτόν έχει ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική όσο υπάρχει τέλμα στα εσωτερικά ζητήματα που θα μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν. Υπάρχει μεγαλύτερη ασυνέπεια λοιπόν και θα υπάρχουν και μεγαλύτεροι κραδασμοί. Ας δούμε την ε, οπισθοχώρηση ε, των ΙΠΑ λόγω χάρη προς την ΠΕΣΚΟ το τελευταίο μήνα η κυβέρνηση Τραμπ δεν ανησυχεί όπως γινόταν παραδοσιακά με τις αμερικανικές κυβερνήσεις στη δεκαετία ότι τα σχέδια άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να την κάνουν ένα στρατηγικό αντεγωνιστή προς, την, ε, προς τη ΣΥΠΑ σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Δεν, δεν ανησυχεί καν στατηγικά ο κ. Τραμπ περισσότερο ε, τον ενδιαφέρει η εμπορική διάσταση της ΠΕΣΚΟ, ότι το αμυντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί τελικά να ε, κάνει διάκριση κατά των Αμερικανικών εταιριών άμυνας. Και αυτό πάλι έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με το εμπόριο παρά με την στρατηγική ε, που θα μπορούσε να έχει καταρτήσει. Μετά, το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στι διαπραγματεύσει παρά στη στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει σοβαρά την διαρκή επικέντρωση του Τραμπ στις διαπραγματεύσεις τις ίδιες. Εκείνος ασχολείται με συναλλαγές από τις οποίες το μεγαλύτερο όφελος για την πλευρά του. Μιλάμε για το ίδιο ε, όφελος και όχι για μια στρατηγική προσέγγιση. Τον ενδιαφέρει το κέρδος, όχι κοινέ αξίες. Και τον ενδιαφέρουν οι απολαβές του παρόντος, όχι οι νοσταλγικές ε, ανακλήσεις του παρελθόντος αυτό που αρέσει στην κυβέρνηση του Τραμπ είναι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Αυτά με τα κοινά ιδεώδη, τι κοινέ αξίε και τι κοινέ αρχέ δείχνουν δυναμία κατά τη διάρκεια των δημοτεύσεων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε έχουν ε, αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τον Τραμπ, να τον κολακεύσουν και να μπορέσουν στι συναντήσει του να πάρουν μια θετική αντίδραση για να την πάνε πίσω στι χώρε του. Δεν είναι έτσι σε μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Ε, είναι σημαντικό να ξέρει κανεί ότι οι θετικέ τη που θα έχει κάποιο από μία συνάντηση δεν θα μεταφραστεί σε κάποια πολιτική κίνηση, δεν θα τη θυμάται καν ο Τραμπ μετά. Ε, αυτό που πρέπει να θυμάται κανεί είναι η λογιστική αντιμετώπιση του Τραμπ στα πράγματα. Τα βλέπει όλα ω συναλλαγέ, αυτό που ανέφερα προηγουμένω. Και μπορεί κανεί να σκεφτεί ότι αν τον απειλήσει με αντιδασμού ή με αντίπεινα στην περίπτωση του Ιράν, αυτό μπορεί και να τον ταρακουνήσει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες καταλαβαίνω ότι σας δυσκολεύει να πατήσετε πόδι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να βγάλει κανείς άκρη με τον Τραμπ. Επίσης, η γεωπολιτική προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ξεχνάει το πόσο πίεση μπορεί να ασκεί το να βρει άλλους κοινούς ε, κώδικες με άλλες ε, μεγάλες δυνάμεις σε σχέση με την κυβέρνηση του Τραμπ. Πρέπει να κοιτάξετε να έχετε ουσιαστικέ ε, συνεννοήσεις και σχέσεις με τις δυνάμεις οι οποίες απασχολούν την, ε, τη ΣΥΠΑ, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις σας με τη ΣΥΠΑ. Όχι η αντιπαράθεση, η εξισορρόπηση του βάρους των ΗΠΑ. Δεν είναι αυτό ο στόχος. Παρά τις εκεντρικότητες της κυβέρνησης του Τραμπ και του ίδιου του Πρόεδρου, η οικονομική, πολιτιστική και ιδεολογική σχέση, είπα, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι, σημαίνουν ότι θα παραμείνουν στενοί γεωπολιτικοί σύμμαχοι. Αλλά σημαντικό είναι να σκέφτεστε όπως, ότι θέματα όπω η συμφωνία του Ιράν, οι κλιματικέ αλλαγέ, οι, οι δασμοί για το χάλιβα και το αλουμίνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, στη συνεννόηση με άλλου στρατηγικού εταίρου και αυτά να ασκήσουν πίεση για να επέλθει κάποια εξισορρόπηση στι ευρωπαϊκέ ευρωαμερικανικέ σχέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαπύρο για αυτήν την ερμηνεία. Θα υπήρχε και τέταρτος ομιλητής, ο κύριος Κέρεμανς, αλλά δυστυχώς ζητά συγγνώμη δεν μπορούσε να έρθει. Για λόγους υγείας, του ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ο οποίος κάθεται δίπλα μου, ο κύριος Λάγκε. Ε, μπορείτε να μας κάνετε κάποιες ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κύριε Λάγκη, έχετε το λόγο. Δύο λεπτά λέει εδώ, αλλά εσείς κανονίζετε. Μπορείτε να πάρετε το χρόνο του άλλου μιλητή. Σας ευχαριστώ, κυρία Συμπρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονές μας σχετικά με το εμπόριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι σημαντικός εμπορικό εταίρο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τι εισαγωγέ και εξαγωγές. Ε, αυτό βασίζεται και σε απόφαση του ΠΟΕ το 1995. Εκδόθηκε μια σειρά αποφάσεων που αποτελούν ένα λόγο της μεγάλης επιτυχίας αυτής στο εμπόριο. Όπως είπε ο κύριος Γκάρνερ, οι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα υπονομεύουν τους κανόνες ε, της, του ΠΟΕ. Υπάρχει νομοθεσία ψυχροπολεμική του 1962 που σχετίζεται με ε, την ασφάλεια, την οποία αποκαλούνται οι Ηνωμένε Πολιτείε και στην περίπτωση της Κίνας ε, την απόφαση 301 του 1974 και οι δύο αυτοί νόμοι δημιουργήθηκαν πριν τον ΠΟΕ. Ήταν απόλυτα σαφές ότι ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε γνώριζαν το 1996 ότι αυτές οι ε, νομοθεσίες δεν ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες του ΠΟΕ. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά ε, τους ε, διεθνείς κανόνες εμπορίου. Τι γίνεται λοιπόν όσον αφορά τις προοπτικές συνεργασίας. Θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το σύστημα παγκοσμίου εμπορίου. Έχουμε όμως το συγκεκριμένο πρόβλημα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν κάνουν κάτι για, την, για τον διορισμό δικαστών ε, στο σχετικό σώμα και έτσι ο ΠΟΕ μπορεί να μην λειτουργεί πια του χρόνου. Ένα βήμα συνεργασία λοιπόν θα ήταν να διασφαλίσουμε το σύστημα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Δεύτερον, ε, για το λευκό οίκο γιατί ε, επικεντρώ αποτελούν μόνο τα προϊόντα, το εμπόριο προϊόντων έχουμε πλεόνασμα όσον αφορά τις υπηρεσίες. Ε, και νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι που βγαίνουν κερδισμένες από το, τη συμφωνία TRIPS. Εκατομμύρια ε, ε, καταλήγουν στις Ηνωμένε Πολιτείε λόγω διπλωμάτων τεχνιών. 30 δισεκατομμύρια από την Κίνα και μόνο. Γιατί λοιπόν επικεντρώνονται οι Ηνωμένε Πολιτείε αποκλειστικά στο εμπόριο αγαθών. και γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν εξετάζουν τη συνολική εικόνα του εμπορίου. Τρίτον, όπως ανέφερε και ο κύριος Γκάρτνερ, ε, δεν ε, ενδείχνεται να ε, διαπραγματεύεται κανείς εμπορική συμφωνία υποπίεση. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι μέτρα θα ήταν χρήσιμα για την καλύτερη αλληλοκατανόηση στο μέλλον. Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να επιτραπεί η πρόσβαση στην αγορά, να δημιουργηθεί σχετική συμφωνία για την πρόσβαση στην αγορά, η οποία να διασφαλίζει την ισορροπία. Δεν μπορούν δηλαδή από τη μία να μειωθούν τα δασμία από τη μία χωρίς να παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα χωρίς πίεση να βρεθεί μια κοινή προσέγγιση για τέτοιες διαπραγματεύσεις πρόσβασης στην αγορά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λάνιε. Έχω εδώ κατάλογο ομιλητών. 10 ομιλητές έχουμε. 11 μαζί με τον κύριο Τάνοκ. 12. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. 1,5 λεπτό κάθε ομιλητής. Ο κύριος Πέτερλε, παρακαλώ. Ω, μα τι προνόμιο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές για τις αφέστατες και ξεκάθαρες ταράτες κουβέντες τους. Από γενετικής σκοπιάς ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, ε, λίγο πολύ, αλλά η γενετική εδώ δεν έχει καμία σημασία. Ως πολιτική έχουμε συνηθίσει μια κάποια προβλεψιμότητα, προβλεψιμότητα που είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη σταθερότητα. Δεν θα συνεχίσω αυτές τις θεωρητικές δηλώσεις, γιατί η συζήτηση σήμερα είναι συζήτηση για την ίδια μας την προσωπική αντίληψη. Ο κύριος Φων Μάρσαλ μας κατήφθηνε στη στο σωστό προορισμό πιστεύω. Η θετική πλευρά της σημερινής κατάστασης είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να δούμε σήμερα. Δεν μου αρέσουν τα συνθήματα περισσότερη Ευρώπη, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη ένωση στην Ευρώπη, πιο ξεκάθαρες ιδέες και περισσότερη πυγμή και αποφασιστικότητα. Ο κύριος Κάρνερ είπε θα επιβιώσουμε. Ε, ο κύριος Κάρτινερ είπε ότι θα επιβιώσουμε, αλλά το θέμα είναι με τι τίμημα. Και ε, ο κύριος Μάρσφερ ανέφερε τα Δυτικά Βαλκάνια. Είπαμε ότι σύνοδος θα γίνει στη Σόφια για το θέμα αυτό, έχει ξεκινήσει και πρόσφατα έγινε και διάσκεψη στη Βόσινγκτον για τα θέματα αυτά και υψηλού επίπεδου με υψηλούς το ερώτημα είναι θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ ή θα έχουμε ανταγωνισμό για αυτή την ιδιαίτερη και ευαίσθητη ευρωπαϊκή περιοχή. Θυμάμαι όταν είχε πει ο Σιράκ πρώτη Γαλλία και καταλαβαίνω που λέει και ο κύριος Τραμπ ε, η, Αμέρικα, η Αμερική πρώτη. Αλλά δεν είναι η τα αποθυμένα αυτά μεγαλείου που με ενοχλούν ε, είναι η ανάγκη να εργαστούμε μαζί και αυτό που μας λείπει προς στιγμή είναι το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε μαζί. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε βαθύτερο διάλογο και κοινοβουλευτικό και διατλαντικό και ότι θα παίξουμε ε, το ρόλο της ήπιας δύναμης ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο λίγο πιο ε, αποφασιστικό. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερλη. Κυρία Γκόμες, παρακαλώ να παραμείνετε στο όριο μιλία σας. Ένα μισή λεπτό. Ναι, σας ε, ευχαριστούμε που ξανά ήρθατε κύριε Γκάρτνερ, πρέσβευτά Γκάρτνερ. Δεν αναφέρατε αυτό που θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει τον ελέφαντα στην αίθουσα, αυτό που είναι μπροστά μας και δεν το βλέπουμε, τον, ε, τη ρωσική διάσταση, τη Ρωσία την ίδια. Ε, ο κύριος Φων Μάρσαλ, ο καθηγητής Φον Μάρσαλ, δεν ε, πιστεύετε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόβλημα το θέμα της ηγεσία, η, πολιτικής, η απουσία πολιτικής βούλησης, η δυσκολία να επιδείξουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να υπάρξει δράση. Διότι όταν βλέπουμε τις αντιδράσεις ε, και τα διάφορα παρασκηνιακά που έγιναν στην περίπτωση του Τραμπ του ίδιου ή την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Τραμπ, στην υπόθεση της Gazprom, ε, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Κύριε Τάνοκ, είστε επόμενος. Ευχαριστώ πολύ να πω ότι μας είχε λείψει ο πρέσβης Γκάρνερ και τα σοφά του λόγια. Χαίρομαι πολύ που τα λέει πάντοτε ξεκάθαρα και τσουβαλάτα. Εδώ λοιπόν ε, σήμερα τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζω ότι ο διάδοχός του που ανέλαβε θα καταφέρει να έχει επιτρέψει με την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο για την κυβέρνηση Τραμπ δύσκολο να ξέρει κανείς ε, τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι επόμενες πολιτικές ε, επιλογές τους, αλλά σε προηγούμενη ζωή μου και λόγω των όσων έμαθα από αυτή την εμπειρία πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω πολύ καλά την προσωπικότητα του Τραμπ. Το είδαμε με τη Συμφωνία των Παρισίων, το είδαμε με, την, ε, με τους δασμούς, το είδαμε με το Ιράν Βλέπουμε εδώ ε, την αντίδρασή του με τη Βόρεια Κορέα. Ε, δύο μεγάλοι ηγέτες που δεν θέλουν να μιλήσουν ένα στον άλλο. Τώρα με το Ιράν και την ε, συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων αποστέλλονται τώρα τα λανθασμένα μιλήματα. Ε, κακή συμπεριφορά και καμία τιμωρία. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και δεν μας εκπλήσει πρόσφατα. Είχα συζήτηση με έναν από τους παλιούς βουλευτές του UKIP και φαίνεται να υπάρχει επιθυμία μεταξύ λαϊκιστών παντού στον κόσμο να απεμπλέξουν, να καταστρέψουν και να ισοπεδώσουν τον πολυμερισμό. Λες και αυτός είναι ο εχθρός τους. Είναι φοβερό ε, ότι αυτό αντιμετωπίζουν ως ζήτημα την παγκοσμιοποίηση και τη διασύνδεση, την ε, την κυκλοφορία των ανθρώπων, το εμπόριο. Θεωρούν ότι όλα πρέπει να θα πάνε στο πίσω, στο να πατήσουν το κουμπί του πίσω. Ίσως να μην θέλουν να πάνε καν στο 1950, αλλά και στο 1850 αν γίνεται. Ε, φαίνεται πάντως να είναι πολέμοι του πολυμερισμού και να θέλουν τα απολύτως εθνικά κυρίαρχα κράτη. Και για το εμπορικά και την πνευματική διεκτησία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα πέρα από τα εθνικά σύνορα στο εμπόριο. Οτιδήποτε άλλο ξεπερνά τη φαντασία τους. κυρία Σχάκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας την άποψή μου για την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων. Η διατλαντική μου καρδιά ματώνει με αυτή την κατάσταση. Και πέρα από τις πρόσφατες εξελίξεις θα δούμε και μια αλλαγή γενεών που θα επηρεάσει τα μάλλα το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων, το οποίο ε, συνδέεται με τα βιώματα της γενιάς του baby boom οι ομιλητέ το έχουν σκεφτεί καθόλου αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η ιστορία θα αντιδράσει πολύ άσχημα τελικά, γιατί δεν θα μπορούμε συνέχεια να απορροφούμε με επιτυχία όλα αυτά τα σοκ που υφιστάμεθα. Η αμερικανική πλευρά θέλει να είναι ρεαλιστική. Εμείς είμαστε ρεαλιστικοί ή θέλουμε να βλέπουμε κάτι καλό ακόμα και σε όλα τα ε, δεινά. Από πλευράς Ουάσιγκτον. Είναι η τακτική τους το διέρη και βασίλευε στα κρατη να στρέψουν το ένα κράτος μέλος εναντίον του άλλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα όσον αφορά στη σχέση με τη Ρωσία. Με ενδιαφέρει να τοποθετηθείτε με αυτό το πρίσμα. Και τέλος, στην εσωτερική συζήτηση στη ΣΥΠΑ για τους δασμούς, για τους εμπορικούς κανόνες, για την Κίνα, για όλα αυτά τα θέματα, για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται τα σημεία εξισορρόπησης έναντι του Πρόεδρου Τραμπ και των α, μη συνηθισμένων εμπορικών πολιτικών που ακολουθεί ο κ. Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους όσοι μας μίλησαν. Να σας πω μια ιδέα που έχω, την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Και θα ήθελα να μάθω αν κάποιος ομιλητής μπορεί να τη σχολιάσει. Μιλούμε για τη σταθερότητα. Τη σταθερότητα στον κόσμο, η οποία σίγουρα σήμερα απειλείται. Και πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα είναι να ξεφύγουμε από το δικαίωμα άρνηση κυρίας που έχουν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό το δικαίωμα αρνησή, κυρία, στο ΒΕΤΟ είχε νόημα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν αποφασίστηκε άλλωστε. Τώρα όμως είναι κάτι το περασμένο, είναι απλά τροχοπέδι. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί καμία χώρα τον εαυτό της που υφίσταται επιθέσεις, γιατί ένας από αυτούς τους πέντε αποφάσισε να πει όχι ή νιέτ. Άρα, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί αυτό να το θέσει επιτάπητος. Ξέρω ότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο χώρες που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ίσως είναι δύσκολο για αυτές. Αν όμως το πιστεύει ο κύριος Μακρόν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στον κόσμο. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε. Μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Να το θέσουμε σαν θέμα, να καταργηθεί το δικαίωμα άρνηση κυρίας, να το θέσουμε πλέον επιτέλους στη δημόσια συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπίλντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύρια Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και εσάς αγαπητοί ομιλητές. Οι κυράωση εναντίον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο Ιράν είναι πολύ ανησυχητικές γιατί η PSA, η Total είναι μεγάλη επιχειρηματική γαλλική όμιλη που μπορεί να επηρεαστούν και να θυγούν ιδιαιτέρως. Αλλά οι ρωσικές κυρώσεις ήταν αυτές που είχαν τιμωρήσει περισσότερο τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το Τζο Μπάιντον είχε αναγνωρίσει τον Ιανουάριο ότι η Ευρώπη είχε υποχωρήσει στις αμερικανικές πιέσεις και είχε επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ενώ δεν είχε τίποτα να κερδίσει από αυτό. Είναι 10 φορές μεγαλύτερο το ευρωπαϊκό εμπόριο με τη Ρωσία σε σχέση με το εμπόριο με τη ΣΥΠΑ. Η Ρωσία είναι ο τρίτη χώρα οικονομικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι η 20 τρίτη η οικονομική εταίρος της ΕΠΑ για το εμπόριο αγαθών. Είναι θλιβερό το ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιβάλλει νέες κυριαώσεις που τιμωρούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και το Nord Stream 2, όπου ε, αυτό επηρεάζει και το, επίσης ε, τιμωρεί και τους μικρούς Γάλλους παραγωγούς, όπως είναι ε, οι τυροκόμοι, οι οποίοι εκτιμώνται ιδιαίτερα στη Ρωσία. Δηλαδή είναι ένα σημείο ρήξη, τιμωρούνται και οι μικροί και οι, μεγάλοι. Πώς βλέπετε ότι μπορούν να διαμορφωθούν οι διατλαντικές σχέσεις σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. κύριος Καστάλντο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους και προσωπικά πιστεύω ότι εν μέρη θα συμφωνήσω απόλυτα με δύο. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο για τον Τραμπ ότι δεν θέλει να έχει και δεύτερη θητεία να ξανακλαγεί. Και το άλλο είναι ότι έχουμε απέναντί μας ε, μια προσωπικότητα, μια φυσιογνωμία που δεν ακούει παρά ε, τις με πυγμή αντιδράσεις του και σε καμία περίπτωση κάτι που να βασίζεται στον πολυμερισμό. Ε, κάτι που είναι ξεκάθαρα από τις παρουσιάσεις σας και το βλέπουμε και από την Αμερικανική κοινή γνώμη. Η εικόνα που έχουν για τον Τραμπ δεν είναι τόσο αρνητική όσο αυτή που έχουμε από αυτή την όχθη του ωκεανού ή και άλλοι εταίροι στον υπόλοιπο κόσμο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Επειδή από κάθε δυσκολία μπορεί να γεννάται μια ε, ευκαιρία, ουδέν κακό αμυγές καλού και είδαμε με τη συμφωνία των πυρηνικών να υπάρχει και μια σοβαρή ευκαιρία εδώ ίσως ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουμε στους εταίρους μας, τους Ιρανούς συνομιλητές, ότι έχουμε την διάθεση και την αποφασιστικότητα να ε, τηρήσουμε το λόγο μας ως τέλος και να έχουμε μια στρατηγική ατζέντα γεωπολιτική ατζέντα ανεξάρτητη, ακόμη και αν διαφωνούμε με τους φίλους μας στη Ουάσιγκτον. Οπότε, εάν υιοθετούσαμε μια σκληρή γραμμή απέναντι σε ενδεχόμενες ε, δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ και απαντούσαμε με το ίδιο όπλο. Πόσο μακριά πιστεύετε θα πήγαινε ο Τραμπ. Αυτό το πόλεμο θα τον έφτανε στο έσχατο σημείο ή μπορεί και να άκουγε τη φωνή της λογικής και του επιχειρηματικού κόσμου, τον είπα, που έχουν ε, σοβαρή και μεγάλη αγορά, που δεν μπορούν να επιτρέψουν στους εαυτούς τους να τη χάσουν. Ούτε κι εμείς μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να χάσουμε την Αμερικανική. Πόσο μακριά πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει. Ευχαριστούμε κύριος Πάμπριξ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ναι, μπορεί να επικρίνουμε τον ε, Τραμπ μπορεί να γελάμε μαζί του, είναι όμως ε, ε, δημοφιλής σε διάφορες τομείς της κοινωνίας και δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε μπορούμε να τον αλλάξουμε ως άνθρωπο και θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι και θα παραμείνει ο βασικός στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης. Υπό αυτή την προοπτική θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε και βρήκα αρκετά ανησυχητικό αυτό που είπε ο κύριος Σαπύρο, ότι κατά των ΗΠΑ και του Τραμπ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική συνεργασία με την Κίνα ή τη Ρωσία. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά. Νομίζω όμως ότι ε, αυτό ακριβώς θα ήθελαν ο Πούτιν και κάποιοι στην Κίνα, η ηγεσία της Κίνας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί ε, τα συναισθήματα να μας πρόξουν να σκεφτούμε έτσι, αλλά οι Αμερικανοί είναι στρατηγικοί εταίροι των Ευρωπαίων με ή χωρίς τον Τραμπ και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτό που έχει πει εδώ κάποιος άλλος ομιλητής. Η Γερμανία δεν μπορεί πια να κρύβεται πίσω από την ιστορία της, θα πρέπει να πληρώνει την άμυνά της ε, και ε, θα πρέπει επίσης να έχουμε περισσότερη ηγεσία από πλευράς του Μακρόν. Εάν θέλουμε ισχυρή διατλαντική συνεργασία, χρειαζόμαστε εδώ σωστή ηγεσία. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ο κόσμος αλλάζει. Πάει ο παλιός ο κόσμος. Και ο Τραμπ, ο Πούτιν, η Κίνα θέλουν να αλλάξουν το κατεστημένο. Διότι νιώθουν ότι είναι ευνοϊκός ο άνεμος αυτή τη στιγμή. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία τύπου TTIP Light. Ο Τραμπ ίσως κάτι τέτοιο να το ήθελε. Αλλά δεν πρέπει να αναβάλουμε πια τις προσπάθειές μας. Η απάντηση βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριο Παντσέρη. Άλλους έξι ομιλητές έχουμε. Και έτσι θα κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Σας παρακαλώ να ε, τηρήσετε το χρόνο ομιλία σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μάρσαλ, καταλαβαίνω αυτό που νιώθετε, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι τελικά μπορεί να καταλήξουμε ε, η πολιτική δύναμη της Ευρώπης να είναι ασήμαντη απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο τους. Όταν ένας εταίρος θέλει να πλήξει ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με κυρώσεις όσον αφορά το θέμα του Ιράν, αυτό μιλάει από μόνο του. Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν ένας φιλικός διάλογος. Δεν, νομίζω, δεν πιστεύετε ότι η νέα φάση που ξεκίνησε με την κυβέρνηση Τραπ που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες χρειάζεται προσπάθεια από όλους εμάς εδώ στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να επανεξετάσουμε την σχέση αυτή από γεωπολιτικής άποψης. Ευχαριστώ κύριε Σμιρανμούν. Παρακαλώ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές, να τους χαιρετήσω και να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου τον κύριο Κάρνερ, με τον οποίο έχω συζητήσει πάρα πολλές ώρες και έχουμε δουλέψει σε αγαστή συνεργασία. Είναι φυσικοί συνεργάτες μας οι ΗΠΑ. Είναι η στρατηγική σχέση πιο σημαντική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι αποκλίνουν οι θέσεις. Όλο και περισσότερο. Και ως προς την κλιματική αλλαγή και ως προς τη μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Υποδνομεύονται, υποβαθμίζονται οι σχέσεις και μάλλον η Ουάσιγκτον και η νέα διοίκηση, η νέα, ο νέος πρόεδρος, ε, όλο και ε, λιγότερο έχουν σε εκτίμηση την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Brexit δεν έχει συμβάλει σε αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι θεραπευτικό μέσο είναι να διατηρήσουμε την ενότητά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, οξύνεται ο λαϊκισμός παντού, οι ευρωφοβικές απόψεις και αυτά θα επηρεάσουν τις εκλογές του 2019. Θα έχουμε ένα κοινοβούλιο πολύ πιο κατακαιρματισμένο και, κατακαιρματισμένο και μια αδύναμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι προβλέπουν ότι δεν θα είναι τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη στο ύψος των περιστάσεων. Εσείς τι πιστεύετε και ποιο θα είναι και το μέλλον της, ε, του Πρόεδρου Τραμπ. Τι θα γίνει με τις εκλογές του φθινοπόρου. Είναι κάτι που θα έχουμε να κάνουμε τα επόμενα δυόμιση χρόνια ή τα επόμενα εξήμιση και χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και μιλούμε για μια εξωτερική πολιτική κάπως ε, περίεργη. Θεωρείται ότι με τη μεταφορά της πρεσβείας ε, στην Ιερουσαλήμ η λύση για τα δύο κράτη είναι πια ανέφικτη. Ποια είναι η άποψή σας. Τι πιστεύετε για την περαιτέρω αποσταθεροποίηση για τις κυρώσεις της ευρωπαϊκής επιχειρήσης ε, σε σχέση και με το Ιράν. Αυτό το μεγάλο κενό που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το καλύψει. Ποιος θα το καλύψει, η Ρωσία, η Κίνα. Πώς πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο ερώτημα, σοβαρό ερώτημα. Ποια η γνώμη σας για το να δοθεί βραβείο Νόμπελ Ειρήνη στον Ντόναλτ Τραμπ για τη δουλειά που κάνει μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας. Και είναι σοβαρό το ερώτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ρούπιχ. Εμένα θα με ενδιαφέρε να μάθω τι σκέφτεται ο Κιμ Τζον Ουν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ε, τώρα που δεν γίνεται πια σεβαστή συμφωνία με το Ιράν. Τι νόημα έχουν οι διαπραγματεύσεις εάν γνωρίζει κανείς ότι το αποτέλεσμα δεν θα τηρηθεί ε, και μπορεί να καταργηθεί ε, έτσι. δεν βλέπω να υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες σε, και πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο να τηρηθεί η συμφωνία. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Δεύτερο θέμα, ο εμπορικός τομέας. Οι επιχειρήσει, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν στο πλευρό μας. Θέλουν να έχουν εμπόριο, να παραμείνουν δραστήριες και γι' αυτό και το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να προωθηθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα στην Ευρώπη και στην Αμερική για να ενισχύσουμε το αμοιβαίο εμπόριο. Και αντί να επιβάλλουμε κυρώσεις υπό την μορφή δασμών, να χαμηλώσουμε τους δασμούς. Ο Τραμπ από τη μία παρέχει φοροαπαλλαγές, από την άλλη ε, επιβάλλει δασμούς που τελικά θα πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές, ε, ενώ οι επιχειρήσεις δεν είναι πια ανταγωνιστικές. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε με κυρώσεις και με κίνητρα και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρουμπίχ. Euh, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λέει ο κύριος Πάχνιο. Η συζήτησή μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ε, σε μια στιγμή κατά την οποία υπάρχει πλήρης ε, αταξία, σε σημείο παροξισμού. Θα ήταν λάθος να πιστεύει κανείς ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ο τρελός του χωριού. Θα ήταν ένα τεράστιο πολιτικό λάθος. Ένα τεράστιο πολιτικό σφάλμα το οποίο διαπράττει η δημοκρατική ιντελικέντσια της Ευρώπης ή οι τεχνοκράτες της Αμερικής. Όλοι όμως έχουν χάσει ενάντια στο λαϊκισμό που κυριάρχησε πριν από 1,5 χρόνο σε σημείο παροξισμού. Και όπως ο συνάδελφος Καν, και εγώ να αναφερθώ στο Παλαιστινιακό ζήτημα, και όταν ακούμε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη να λέει ότι τελικά το Ισραήλ επέδειξε αυτό συγκράτηση όταν πυροβολούσε με αληθινές σφαίρες και σκότωνε μικρά παιδιά και νέους ανθρώπους με 60 θανάτους και διάφορους εκατοντάδες και χιλιάδες τραυματίες. Αυτή είναι μια λαϊκιστική, εθνικιστική ρητορική και δυστυχώς τη συμμερίζονται αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμερίζονται διάφορες χώρες που είναι φίλιες και σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ βέβαια επαναλαμβάνω προς την, το Παλαιστινιακό ζήτημα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιος είναι ο ρόλος αυτών των χωρών σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και την Αμερικανική κυβέρνηση. Ποιος έχει τα ενία Τίθεται αυτό το ερώτημα και το είπατε και εσείς νωρίτερα, οι Ευρωπαίοι, εμείς, είμαστε ιδιαίτερως διαιρεμένοι, ειδικότερα ως προς το Παλαιστινιακό ζήτημα. Σήμερα το πρωί ήμουν σε μία συνάντηση με τον Πιάβη ο οποίος είναι στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας και μου έλεγε ότι πρέπει να βρούμε άλλες εταιρικές σχέσεις, να διευρύνουμε το κουαρτέτο με την Κίνα, με την Νότια Αφρική, με την Ινδονησία, με την Ινδία. Και θέλω να μάθω και τη δική σας γνώμη από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Κάλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου που βλέπω τον φίλο μας, τον πρέσβη Γκάρνερ εδώ. Και επίσης να τον ε, συγχαρώ και να το ευχηθώ για τα γενέθλιά του. Είναι τα γενέθλιά του σήμερα. Ε, θα ήθελα όμως να συμφωνήσω με αυτό που και ο συνάδελφος Πέτερλε. Γενετικός ανήκουμε στην ίδια οικογένεια και από τη μια και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και γενετικός και πολιτικός και από πλευράς αξιών. Η χημεία μας είναι τέτοια. Είναι καλό αυτό να το θυμόμαστε συνέχεια. Έχουμε ίσως διαφορές στρατηγικής. Πάντοτε τις είχαμε. Όμως, είναι στρατηγική η σχέση μας, στρατηγική σημασία. Δεν έχουμε καμία εναλλακτική σε αυτό. Να μην μπερδευόμαστε λοιπόν και οδηγούμαστε σε σύγχυση λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του Πρόεδρου Τραμπ. Εάν ασκήσουμε πίεση στην τωρινή Αμερικανική κυβέρνηση, επιζητώντας νέες συμμαχίες με την Κίνα ή τη Ρωσία, όχι μόνο θα φανούμε ότι προσπαθούμε να παραπλανήσουμε, αλλά και θα φανούμε και ανεύθυνοι, εντελώς επικίνδυνοι. Πριν από δύο μέρες ακούσαμε τον Τότεμπερκ να λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε συνεχίζουν να είναι ταγμένες στο ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο με λόγια αλλά και με δράσεις. Άκρισαν την παρουσία του στην Ευρώπη, ε, προσέφεραν περισσότερα στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό και την οικονομική τους συνεισφορά ε, στην Ευρωπαϊκή ε, Ασπίδα Ασφαλείας. Είναι σημαντικό λοιπόν να το θυμόμαστε και να το εκτιμούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλα. Η κυρία Ροντρίγκης Πενιέρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Κάρνερ. Καλώς ορίσατε και πάλι. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και χαίρομαι διότι κατέστη δυνατόν να την έχουμε αυτή τη συζήτηση. Το χειρότερο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας είναι ένας άνθρωπος που ονομάζεται Donald Trump. Και ήταν μια στρατηγική. Μέχρι τώρα έχει, υποσχεθεί, έχει εκπληρώσει όλα όσα έχει υποσχεθεί προεκλογικά. Έχει μεταφέρει την πρεσβεία στην Παλαιστίνη, έχει αποσυρθεί από τη Συμφωνία για το Κλίμα, από την ΑΦΤΑ, από διάφορα πράγματα. Μας εξέπληξε και η απόσυρσή του από την συμφωνία για το Ιράν. Πραγματικά πιστεύετε ότι λειτουργεί άνευ στρατηγική. Εγώ δεν το πιστεύω. Η σύμμαχή του είναι το Ισραήλ και η Σαδική Αραβία και ο εχθρός του είναι το Ιράν. Και ε, για το Ιράν εχθρός είναι η ΙΠΑ. Το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο. Δεν το είπε στην προεκλογική του εκστρατεία, αλλά το κάνει. Και αμφισβητεί την ε, πολυμερή εξισορρόπηση και τα πολλαπλά κέντρα επιρροής. Δεν θέλει να λύνονται οι συγκρούσεις με το διάλογο και με τη διαπραγμάτευση. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού, γιατί εγώ πιστεύω το εξής. Μήπως πίσω από τον Ντόναλτ Τραμπ κρύβονται συμφέροντα που θέλουν τη διεθνή παγκόσμια αστάθεια. Ποιες είναι οι προσδοκίες για τα εκλογικά αποτελέσματα σε πρόθεσμη βάση το Νοέμβριο. Αν οι προσδοκίες είναι ευνοϊκές, τότε θα προχωρήσει με αυτή την άγουσα. Ποια αίσθηση έχει ο Αμερικανικός λαός για τις απαντήσεις που δίνει ο Ντόναλτ Τραμπ σε διεθνείς προκλήσεις και στην παγκόσμια αστάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράγκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ζούμε σε καιρούς μεγάλης οικονομικής αλληλεξάρτησης και μεγάλου πολιτικού κατακαιρματισμού. Και είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς τη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα και να μαντέψει τι θα συμβεί στο μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα μειωθεί ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050, θα είμαστε το 6% του παγκοσμίου πληθυσμού, οι δύο Αμερικές το ίδιο, Βόρεια και Νότια Αμερική. Δηλαδή αυτό το οποίο θεωρεί το Δύση παλιά θα είναι κάτω από το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και αυτή η δημογραφική γύρανση συνεπάγεται και οικονομική φθορά και συρρήκνωση. Είδαμε την άνοδο της Κίνας, διαφόρων άλλων χωρών. Ε, συνεπάγεται αυτό πολύ σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Έχουμε ανάδυση νέων δυνάμεων πολιτικών, νέων χωρών που δεν συμμεριζονται τις απόψεις μας στον τρόπο με τον οποίο εμείς επιλύουμε τις συγκρούσεις. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πολύ απλό. Είμαστε πολύ μακριά από την εποχή όπου το, από το 1870 μέχρι το 1903 ή 30 ήμασταν το 20% του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά και στη δεκαετία του 80 στον 20ο αιώνα είχαμε πολύ μεγάλο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε επιρροή στο πεπρωμένο του παγκοσμίου γίγνεσθε ή θα υπάρξει πολιτική, οικονομική, κοινωνική και θεσμική αλλαγή στη διακυβέρνηση του κόσμου με, την, με τον ε, πρόεδρο Τραμπ. Ε, θα έχουμε δηλαδή κοσμογονικέ αλλαγέ και θα αλλάξει η παγκόσμια τάξη των πραγμάτων έτσι όπω την γνωρίσαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και εγώ κάτι. Μετά την προεκλογική εκστρατεία, γιατί κάποια πράγματα τα είδαμε στην προεκλογική εκστρατεία, ήταν ε, χάρη εκστρατεία. Τώρα ο κύριο Τραμπ εφαρμόζει τι πολιτικέ του και παρόλα αυτά, την εταιρική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ θέλουμε να, τις, ε, να τη διατηρήσουμε, είναι προφανές. Στη συζήτηση όμως επίσης προφανές κατέστη ότι χρειάζεται και άλλη συζήτηση. Όλοι έχουν κάτι να πούν και πάντα θα υπάρχει κάτι να πούμε. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να απαντηθούν διεξοδικά σήμερα. Θα κάνω όμως το εξή. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Μπροκ ε, ως τελευταίο μιλητή που είναι ο εισηγητής μας. Έχουμε στις τέσσερις. Οπότε δίνω δύο λεπτά στον καθένα από τους ομιλητές. Είναι περισσότερα από αρκετά, έτσι. Ωραία, τέσσερα λεπτά στον καθένα σας. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γκάρντνερ. δεν ήθελα να κάνω τίποτα διαφορετικό στα γενέθλιά μου. Ήθελα να βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας. Να με προσκαλέσετε και το χρόνο λοιπόν. Ήταν πολλά τα ενδιαφέροντα σχόλια, θα επικεντρωθώ σε μερικά μόνο. Κοιτάξτε, το Νόμπελ Ειρήνη ονομάστηκε Νόμπελ Ειρήνη. Υπάρχει η λέξη Ειρήνη για κάποιο λόγο. Δεν ονομάστηκε Νόμπελ Πολέμου, ούτε Νόμπελ Αποσταθεροποίηση. Πολλοί ομιλητέ είπαν ότι είναι σημαντικό να δουλέψουμε από κοινού για πολλά θέματα. Ε, και Σίμπερτ ε, ανέφερε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Ε, στο εμπόριο, παρά τι διαφωνίε μα, κάποιε διαφωνίε για το TTIP. Είναι τόσο σημαντικό μελλοντικό εργοτάξιο ή τα αγαθά. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα αγαθά απλοϊκή μου απάντηση είναι ότι αυτό το επιλέγει ο Τραμπ γιατί μάλλον αφορά τους πληροφόρους του ε, και τους βιομηχανούς. Βεβαίως η άειλη ε, εμπορική διάσταση μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα, αλλά δεν έχει κανένα οικονομικό νόημα να επικεντρώνεται τόσο πολύ στα αγαθά, αλλά αρέσει στους προφόρους του. Γιατί να αποσυρθούμε και να, ε, να αποχωρήσουμε από την Συμφωνία των Παρισιών. Γιατί πολλές θέσεις εργασίας που έχουν σχέση με τα ορεκτά καύσιμα και όχι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρέσουν στην ε, βάση του, στους ψηφοφόρους του. Επίσης, για το τίτι που είναι πολύ ισχνό και δεν ασχολείται με τίποτα πέρα από την πρόσβαση στην αγορά. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι οι δημόσιες προμήθειες έχουν γίνει τώρα πολύ δύσκολο θέμα σε σχέση με την προηγούμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Ήταν ήδη δύσκολο στην αρχή των διαπραγματεύσεων, πόσο μάλλον με τον Τραμπ, οι θαλάσσιες μεταφορέ το ίδιο. Δεν βλέπω λοιπόν η πρόσβαση της αγοράς να διευκολύνεται για την ε, μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένε προτάσει για να λειτουργήσει καλύτερα ο ΠΟΕ και αυτό το έχει υποσχεθεί η Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Μόνο λέει ότι θα διορίσει τα δικά τη μέλη, αυτά που αρέσουν και θα ε, παρεμποδίσει ολόκληρο το σύστημα. Ο ΠΟΕ ε, λέει ξεκίνησε για να υπάρξει συμφωνία με την Κίνα. Ωραία, πείτε μα λοιπόν συγκεκριμένα με προτάσει επιτάπητο πώ να λειτουργήσει καλύτερα ο ΠΟΕ, αλλά δεν το κάνουν. Επίσης, πολύ γρήγορα, υπάρχει μια ολόκληρη πλειάδα θεμάτων που θα πρέπει να τις μελετήσουμε από κοινού. Ανέφερα μερικές επιδοτήσεις, η πνευματική ιδιοκτησία, η μεταφορά αυτής, η πρόσβαση σε αγορές των χωρών. Αυτά είναι πράγματα που θα μας απασχολήσουν και από κυβερνητικές απόψεις έχουμε κοινά συμφέροντα και για την επιβολή του νόμου ε, εδώ δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είδατε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ηλεκτρονικά υποδεικτικά στοιχεία. Κάτι παρόμοιο με αυτό που επιδιώκουμε στις ΗΠΑ με το νόμο Cloud, όπως ονομάστηκε, το Cloud Act. Εδώ λοιπόν καλό θα ήταν να συμβαδίσουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αποδοχή αποδεκτικών στοιχείων για σοβαρά πανικά εγκλήματα. Και τελευταία κουβέντα. Να επικεντρεθούμε στα θετικά, διότι είδαμε ο πολιτικός κόσμος των ΗΠΑ να ανταποκρίνεται. Δείτε τι γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το τι γίνεται με τα post του Los Angeles Times, ας πούμε, ε, ή με τους νέους που πάνε να ψηφίσουν μαζικά στις επόμενες εκλογές. Τι γίνεται με τους δικαστές μας ε, και το πώς αντισταθμίζουν την πολιτική εξουσία ως θεματοφύλακες του συντάγματο. Είναι νομίζω ένα ε, ξύπνημα όλο αυτό που συμβαίνει, μια ευκαιρία για ξύπνημα και θα πρέπει να το βλέπουμε το θέμα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστούμε κύριε Γκάρντνερ, κύριε Φον Μάρσαλ. Thank Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Νιώθω ακόμα εδώ, πώς να το πω, ότι ο κόσμος θέλει να λιδωρήσει τον Τραμπ, να παραπονεθεί για τον Τραμπ. Ναι, από συναισθηματικής πλευρά αυτό ε, είναι κατανόητο, αλλά αυτό δεν βοηθάει μετά από 1,5 χρόνο. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε στρατηγικά και πώς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Αυτό είναι σημαντικό για μένα, να ξεφύγουμε από ε, τις κοροϊδίες και τα παράπονα ε, στο να πάρουμε στα σοβαρά τα δικά μας συμφέροντα. Ε, ναι, πράγματι σέβεται ε, την, ε, όταν ασκείται πίεση από την αντίθετη πλευρά, έτσι λειτουργεί ο Τραμπ. Και εάν διαπιστώσετε ότι σήμερα σε σχέση με την πρώτη φορά που συνάντησε την κυρία Μέρκελ, σίγουρα τη σέβεται περισσότερο, αλλά δεν πρέπει να αγωνιστεί κανείς αν δεν πρόκειται να κερδίσει. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία TTIP Light. Ναι, θα μπορούσε η ευρωπαϊκή πλευρά να προτείνει απαλλαγή από δασμού. Έχουμε υψηλότερου δασμού από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει δίκιο σε αυτό ο Τραμπ. Αλλά αυτό δεν ε, θα αρκέσει, διότι ο κύριος Ρο έκανε απόλυτα σαφές ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί να μετακινηθεί, να αλλάξει θέση όσον αφορά τα μη δασμολογικά θέματα. προστασία του καταναλωτή, γεωργία, αυτά είναι θέματα που τους ενδιαφέρουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα μέχρι την 1η Ιουνίου. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Πολλοί ρώτησαν σχετικά με τα μέσα της θητείας. Εάν, διαπιστώσετε, εάν παρακολουθείτε τις εξελίξεις θα δείτε ότι 6 ε, με 7% είναι το προβάδισμα των δημοκρατών. Εάν όμως αυτό κανείς το μετατρέψει σε έδρες, ε, το επίπεδο είναι λίγο πολύ το ίδιο. Είναι λοιπόν ανοιχτό ερώτημα το αν μπορεί, μπορούν οι δημοκρατικοί να ξανακερδίσουν ε, την Βουλή των Αντιπροσώπων ε, και όσον αφορά τη Γερουσία είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών ε, θα έχει σημαντικές ε, ψυχολογικές επιπτώσεις. Εάν οι δημοκράτες δεν μπορέσουν να ξανακερδίσουν την Βουλή των Αντιπροσώπων, ε, θα βρεθούν στην έρημο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που θα ευνοήσει την επανεκλογή του Τραμπ. Εάν όμως ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τότε θα έχουμε δύο χρόνια πολιτική πολιτικών ε, μπλοκάζ στις Ηνωμένε Πολιτείε, διότι δεν θα επιτρέψουν να περάσει καμία πρόταση. Άκουσα να λέγεται ότι ο Τραμπ είναι το χειρότερο πράγμα που μας συνέβη τα τελευταία χρόνια. Όχι, εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλά χειρότερα πράγματα οι έλεγχοι και τα αντισταθμιστικά μέτρα λειτουργούν καλά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μπορεί να μην μα αρέσει το στυλ του, το ύφο του, μπορεί να μα αρέσουν οι απόψει του, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, συνεχίζουν να αποτελούν δημοκρατία και να είναι ο πιο σημαντικό μας εταίρο. Και σίγουρα δεν αποτελεί ε, θεμητή λύση η Κίνα ή η Ρωσία. Επίσης, ε, ναι, σκέφτομαι το θέμα που είπατε, υπάρχουν νέες γενιές που δεν έχουν ζήσει τον ψυχρό πόλεμο. Οπότε δεν βλέπουν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης. Ε, από την άλλη βλέπω ότι στην Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ε, δεν ε, εντυπωσιάζονται οι νέοι από την μόδα, από την Ινδία, την ε, μουσική της Κίνας ή τα νέα από την Κορέα. Η λαϊκή κουλτούρα της Αμερικής τους έχει επηρεάσει και με αυτό μπορούμε να εργαστούμε. Αυτό συχνά ε, συνδέεται και με αρνητικό πολιτικό αίσθημα απέναντι στι ΗΠΑ. Νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ κύριε Σαπύρο. Οι τελευταίε σα παρατηρήσει. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα τέθηκαν. Δεν ε, θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα, αλλά ελπίζω να συνεχιστεί η συζήτησή μα πάνω στα θέματα αυτά. Αρκετοί νομίζω ανέφεραν ότι το θέμα δεν είναι να κοροϊδεύουμε τον Τραμπ, είναι να προτείνουμε λύσεις και απαντήσεις στα όσα κάνει. Ναι, μπορούμε και να το κοροϊδεύουμε, αλλά αυτό δεν αποκλείει και πιο επικοδομητικές λύσεις. Το θέμα είναι, αν το καλοσκεφτείτε, διότι αρκετοί ανέφεραν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο, ο βασικός εταίρος ε, της Ευρώπης, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ουσία της δουλειάς μας είναι να διατηρήσουμε την ε, φιλελεύθερη τάξη και την ε, διατλαντική ε, σχέση. Ναι, αυτό είναι ο στόχος, αλλά πώς θα γίνει αυτό, αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δεχτούμε, να ομολογήσουμε ότι τον Τραμπ δεν τον νοιάζουν αυτά τα πράγματα, δεν τον νοιάζει η, η τάξη, τα, η ελευθερία. Ε, και εμείς μπορεί να μιλάμε εδώ πέρα για ε, κοινέ αξίες και κοινά συμφέροντα. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε λοιπόν τη σχέση αυτή παρά τα τέσσερα ή 8 ή 12 χρόνια με τον Τραμπ πρόεδρο, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να του ασκήσουμε αρκετή πίεση, ώστε να είναι σημαντικό για τις Ηνωμένε Πολιτείε να παραμείνουν εντός αυτής της τάξης, εντός αυτής της διατλαντικής σχέσης και αυτό θα απαιτήσει την εξέβρεση άλλων τρόπων άσκησης πίεσης. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, εάν πούμε απλά ωραία έχουμε τους ε, διάφορους ε, τρόπους ελέγχου και, ε, και εξισορρόπησης, τότε ο, ο, ο Τραμπ ε, θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που θα πρέπει να βρούμε. Και προφανώς η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία δεν αποτελούν υποκατάστατο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν δικά τους προβλήματα όσον αφορά ε, ε, την ελευθερία και τις ευρωπαϊκές αξίες. Όσον αφορά όμως συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα θέματα τακτικής, ε, θα είναι χρήσιμο να φροντίσουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε να παραμείνουν στο κέντρο, στο, που είναι, αυτό που μας ενδιαφέρει δηλαδή ιδιαίτερα είναι η διατλαντική σχέση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαπύρο. Και τώρα φτάνουμε στον κύριο Μπροκ, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής μας, που είναι, προ... που είναι εισηγητής, συγγνώμη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. No, We don't connect. Okay. The floor is yours. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τζέρεμι, ε, χρόνια σου πολλά και από μένα. Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις σημαντικές τους παρατηρήσεις, τις οποίες αξίζει να σκεφτούμε. Αξίζει να αναρωτηθούμε σχετικά με τα όσα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης. Στο σχέδιο έκθεσής μου ε, παρατήρησα ότι ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθώ τις εξελίξεις. γράφω έκθεση, αλλά μέχρι να μεταφραστεί ε, η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ναι, μας εκνευρίζει η πολιτική του Τραμπ σε κάποια θέματα. Ε, είναι σοφή η στάση του στο θέμα του Ιράν. Έχουμε το θέμα των εμπορικών σχέσεων. Έχουμε το θέμα ότι δεν τηρούνται οι κανόνες, οι πολυμορείς κανόνες του εμπορίου. επίσης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι θέλουμε δίκαιο, δίκαιες εμπορικές σχέσεις και εγώ αποφασίζω ότι είναι αυτό. Και όλοι τον υποστηρίζουν σε αυτό. Ανακοινώνει Ε, την ε, απόσυρση του από τους πολυμερούς κανόνες εμπορίου. και φροντίζει όλα να γίνονται προς όφελος των Πολιτειών ε, Αυτό είναι το βασικό του θέμα, με όλη την αβεβαιότητα που προκαλεί αυτό. Κάποιος είπε ότι θα πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε να αντισταθούμε, αλλά μέχρι πότε θα μπορούμε να αντιστεκόμαστε. Διαπιστώνω ότι οι γερμανικές ενώσεις επιχειρήσεων είπαν ότι όχι δεν θέλουμε αντισταθμιστικές κυρώσεις, ενώ διαπραγματευόταν ο Μακρόν και η Μέρκελ στη Ουάσιγκτον. Ε, τότε τι κάνουμε. Δεν αναγνωρίζει διεθνείς κανόνες λοιπόν ο Τραμπ και μάλιστα εφαρμόζει αυτό που έχουν κάνει και στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξοεδαφικά μέτρα. Έχουμε απόφαση της Γερουσίας για το Nord Stream 2. ό,τι απόφαση ληφθεί για τον Nord Stream 2 δεν θα πρέπει να γίνει ε, με βάση ε, εξωεδαφικά μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν διαπραγματεύεται με τους εταίρους, ε, τους ανακοινώνει τι πρέπει να κάνουν, αλλιώς θα τιμωρηθούν. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Βερολίνο μία ώρα αφότου ε, παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του, ε, ανακοίνωσε ότι θα πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να αποχωρήσουν από την ε, συμφωνία με το Ιράν αμέσως. Αυτό προκαλεί ανησυχία. Πώς λοιπόν θα χειριστούμε αυτήν την εταιρική σχέση. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι είναι ο σημαντικότερος εταίρος μας. Ναι, η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά έχει αξιοπιστία μια εταιρική σχέση όταν, ο, όταν ένας εταίρος δεν γνωρίζει καθόλου τι θα συμβεί αύριο. Όταν δεν υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι πάντα ισχύει το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι θέματα που οδηγούν σε αβεβαιότητα. Οι Αμερικανοί, μετά το θέμα με την Ουκρανία, βοήθησαν μέσω του ΝΑΤΟ, αλλά ο Ομπάμα είχε λάβει τη σχετική απόφαση, όχι ο Τραμπ. Ο Ομπάμα τα αποφάσισε όλα αυτά. Βρέθηκε στην Ασία μια αποστολή της ΑΦΕΤ, όπου διαπιστώσαμε την ανησυχία των Ιαπώνων. Φοβούνται ότι θα υπάρξει συμφωνία αξί Τραμπ Ε, και ο κλασικός εταίρος ε, των ΗΠΑ, η Ιαπωνία, δεν ε, νιώθει καθόλου ασφαλής. Η Συμφωνία του Ειρηνικού στόχο είχε να προστατεύσει τους συμβαλωμένους από την Κίνα. Η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και άλλες τέτοιες χώρες τελικά αναρωτιούνται μήπως θα πρέπει να έχουμε συμφωνία με τους Κινέζους τη στιγμή που ε, δεν είναι σίγουρο ότι θα μας προστατεύσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλάζει λοιπόν η αρχιτεκτονική της ασφάλειας στον κόσμο. Η Αμερική εγκαταλείπει την θέση του παράγοντα που προστατεύει, που διασφαλίζει την ασφάλεια στον κόσμο. Σε τέσσερις εβδομάδες θέλουμε να κλώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία αλλά ε, εάν ε, δεν υπάρχει αυτή η στρατιωτική διάσταση, το κενό μόνο εν μέρη θα συμπληρωθεί. Και έτσι, με την ε, ανασφάλεια στην Ασία, δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε σε άλλα προβλήματα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πλήρη συνείδηση των κινδύνων. Οι Αμερικανοί υπόθηκε έχουν εγκαταλείψει κάθε στρατηγικό προβληματισμό και σκέφτονται με βάση συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες διότι από οικονομικής πλευράς ε, και οι δεσμοί για τον Χάλιβα δεν έχουν κανένα νόημα. Εγκαταλείπουν λοιπόν κάθε στρατηγική. Οι Ρώσοι έχουν στρατηγική, δεν έχουν όμως μέσα να την εφαρμόσουν, διότι είναι φτωχή χώρα. Οι Ευρωπαίοι έχουν τα μέσα, αλλά καμία στρατηγική. Μόνο οι Κινέζοι έχουν και στρατηγική και πόρους. Εάν λοιπόν τώρα διαλυθεί η Δύση, εάν δεν υπάρχει κοινή δυτική στρατηγική, και το TTIP είχε στόχο όχι μόνο την απαλλαγή από δασμούς, αλλά και μια ε, παγκόσμια στρατηγική με βάση την οικονομία. Το θέμα δηλαδή δεν ήταν μόνο οι δασμοί. Είχε και άλλη διάσταση και μια ενδεχόμενη συμφωνία TTIP Lite. θα μπορούσε να μας βγάλει από την κρίση αυτή, δεν έχει όμως στρατηγική διάσταση. Περνάω όμως γρήγορα στο βασικό νόημα. Ισχύει ότι είμαστε εταίροι και ότι η ύπαρξή μας εξαρτάται από την εταιρική αυτή σχέση. Θα έπρεπε αυτό να είναι σαφές. Οι Αμερικανοί έχουν ε, μεγάλο ε, εμπορικό πλεόνασμα, έχουν όμως ε, και τεράστιο εξωτερικό χρέος. Οι Αμερικανοί μαζί με τους Ιάπωνες, τους Κινέζους και τους Ευρωπαίους έχουν συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια χρέος. Διαπιστώνουμε επίσης ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες διότι αντισταθμίζουμε ένα στις αδυναμίες του άλλου. Μαζί είμαστε ο πιο σημαντικός, ο πιο ισχυρός παράγοντας στον κόσμο, οικονομικά και πολιτικά. Αυτό σημαίνει όμως ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουν. Και δεν αναφέρομαι στα 2% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Δεν θέλω να σας διακόψω, λέει η Πρόεδρος, αλλά... Το επόμενο θέμα είναι η έκθεσή σας. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, λέει ο κύριος Σπρόκ. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε πιο ισχυρή θέση, όχι όσον αφορά το 2%. Το, με το 2% μπορεί να δημιουργήσουμε λάθος δομές, να σπαταλήσουμε πάλι τους πόρους και να μην έχουμε τελικά μια ε, κοινή πολιτική ασφαλείας. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις δομές, διότι εάν διατηρήσουμε τις παλιές δομές, και αν δεν έχουν όλοι την απαραίτητη βούληση και με την έλλειψη αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών θα χρηματοδοτήσουμε τελικά την ανοικοδόμηση της Συρίας ε, την οποία δεν καταφέραν οι Ρώσοι και που δεν θέλει ο Ασάντ και τελικά θα καταλήξουμε να κάνουμε όλα αυτά που παραλείπει να κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Μακρόν και άλλοι είπαν ότι βασική προϋπόθεση είναι η Ευρώπη να είναι ισχυρή και να είναι ισχυρός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Σε αυτή τη φάση να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η ερμηνεία και ανάλυση. Και η συζήτηση αυτή προφανώς πρέπει να συνεχιστεί, διότι πρέπει λίγο να αποσαφηνίσουμε τις σχέσεις μας και να δούμε ποιο είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε Γκάρνερ, κύριε Σαπύρο και κύριε Φων Μάρσαλ για την ε, παρουσία σας. Και ελπίζω θα συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε αμέσως για το επόμενο σημείο. Είναι η έκθεση του κυρίου Μπροκ, κύριε Μπροκ. Είναι η δική σας έκθεση